διάθεση των καταναλωτών και τελευταίο εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τελευταίο αλλά σημαντικό. Και εγώ σε ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για την ε, ε, πολιτική κατανάλωση έχει ολοκληρωθεί. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι τα τυχερά παιχνίδια τη απευθεία σύνδεση στην εσωτερική αγορά. Πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Κρόιτσμαν, στον οποίο θα δώσω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές που, για την εξαίρετη πραγματικά συνεργασία τους μαζί μου που έδωσαν δυνατότητα να έρθει φως αυτή η έκθεση και υπερψηφίστηκε με 30 ψήφους υπέρ. Τα τυχερά παιχνίδια ε, βρίσκονται σε μια διασυνοριακή αγορά οι καταναλωτές μπορούν να παίξουν στο διαδίκτυο ε, παιχνίδια τα οποία δεν υπόκειται σε καμία ρύθμιση ή τα οποία επιτρέπονται σε άλλες χώρες όπου ισχύουν άλλες διατάξεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ορισμένες χώρες μέλη να μην έχουν επαρκή προστασία για τους δικούς τους καταναλωτές. Τα παιδιά και οι νέοι τα... Ε, γίνονται εύκολα θύματα εθισμού πολύ συχνά υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός από το εξωτερικό και κάθε χρόνο χάνονται εκατομμύρια ευρώ έσοδα από φορολογία. Είναι σημαντικό θέμα η νομική ασφάλεια όσον αφορά τα χειροπαιχνίδια στην εσωτερική αγορά. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ για την αδειοδότηση. Γι' αυτό θα πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση κατά πόσο οι πρακτικέ των χωρών μελών είναι συμβατέ με το ευρωπαϊκό δίκαιο το ε, υπάρχουσα νομική βεβαιότητα, η νομική αβεβαιότητα ε, αποδεικνύεται από πάρα πολλές ε, παραβιάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει κατεπηγόντως να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα οι χώρες μέλη θα πρέπει να θέσουν το ζήτημα αυτό στο επίκεντρο της προσοχής τους και θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αλλά αυτό δεν επαρκεί για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Επιπλέον θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μελλοντικά να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ζήτησε η Επιτροπή μας με πλατιά πλειοψηφία θα πρέπει να εξεταστεί μια ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή, η οποία να θέτει αλλάξει προδιαγραφέ για την προστασία των ανηλίκων και την καταπολέμηση τη εγκληματικότητα στον τομέα αυτών των τυχερών παιχνιδιών σε απευθεία σύνδεση. Ε, Βεβαίω ισχύει η αρχή τη επικορικότητα. Οι χώρε ε, μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν την κυριαρχία του όσον αφορά τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και να το ρυθμίσουν αυτόνομα. Ωστόσο, θα ε, ε, ε, σε συνάρτηση με τι αφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες. Κρατικά μονοπόλια είναι μόνο επιτρεπτά εφόσον είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα να εδραιώνει το κρατικό της μενοπόλιο με το επιχείρημα της προστασίας του καταναλωτών και από την άλλη να προάγει έντονα διαφήμιση για τυχερά παιχνίδια. Για παράδειγμα, η Γερμανία, όπου έχουμε ένα κρατικό μονοπόλιο για το λότο, αλλά από την άλλη υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, διαφημίσεις και δίδουν ε, ερεθίσματα στους παίκτες να επενδύουν εκεί τα χρήματά τους. Για να βαφηθούν τέτοιου είδους περιπτώσει μελλοντικά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατυπώσει ενιαίες προδιαγραφές ποιότητας για κρατικέ αντιδοτήσεις εάν μια χώρα αποφασίσει ένα κρατικό σύστημα αδειοδότησης θα πρέπει να φροντίσει για την διαφάνεια και την ισότητα. Θα πρέπει όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών ε, στον χώρο τεχερών παιχνιδιών που πληρούν τις προϋποθέσεις να έχουν την δυνατότητα υποβολής ε, αιτήματος για αδειοδότηση. Ταυτόχρονα θα πρέπει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ενισχυθούν ούτως ώστε να υπάρξει μια ενισχυμένη συνεργασία. Πέρα από αυτό θα πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τις χρηματικές ροές μεταξύ παράνομων παρόχων και να απαγορεύσει τις παράνομες δραστηριότητες του. Για παράδειγμα αυτό θα μπορούσε να συμβεί με το κάθε, να υποβάλει κάθε χώρα ένα κατάλογο με τους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών και οι τράπεζες, οι πιστοτικά ιδρύματα θα πρέπει να επιτρέπουν χρηματικές συναλλαγές μόνο με αυτούς τους αδεδοτημένους παρόχους. Το να, ε, το παρεμποδιστεί η εμπλοκή στο ίντερνετ ε, δεν μας βρίσκει σύμφωνο σε εμάς τους ε, φιλελεύθερους. Από τα μέτρα τα οποία διατυπώνει η έκθεση θα επωφεληθούν οι πάροχοι υπηρεσιών οι ρυθμιστικές αρχές και οι καταναλωτές. Παρ' όλα αυτά η Επιτροπή χρειάζεται την πλήρη κάλυψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτω ώστε να μπορεί να υποβάλει τι αναγκαίε πρωτοβουλίε. Γι' αυτό ελπίζω στην ε, αυριανή ψηφοφορία να υπάρξει πλατιά υπερψήφιση τη έκθεση με μια εντολή προ την Επιτροπή. Ο Επίτροπος, ε, ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Μπαρνιέ, παρακαλώ να αναλάβετε αυτό το έργο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρόιτσμαν. τώρα στο πλαίσιο διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε την κυρία Ιώτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση και η πράσινη βίβλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστούν σωστά βήματα μετά από ε, σειρά ετών συζήτησης για να ρυθμίσουμε κάτι που δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Δηλαδή τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια που είναι διασυνοριακά, όχι μόνο ανάμεσα δηλαδή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς όμως θα προστατεύσουμε τους καταναλωτές κατά της απάτης, ε, πώς να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρημάτων, πώς να προστατεύσουμε τους ανηλίκους από τα τυχερά παιχνίδια. Όλα αυτά σε επίπεδο Λοιπόν, ε, σε αυτό το στάδιο είμαι υπέρ ε, των ε, εθνικών πολιτικών. Δεν θα πρέπει όμως η αρχή της επικροϊκότητας να εμποδίσει την εντονότερη συνεργασία για την καταπολέμηση οργανωμένων εγκληματικότητα Στην παράγραφο 20 θα πρέπει, θα πρέπει να τη διαγράψουμε, διότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίνουν τους αποχρόντες λόγους αν πρόκειται να αποκλίνουν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σας ευχαριστούμε, αλλά έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Σας διακόπτουμε, κυρία Έργον Πέρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Βρισκόμαστε ε, μπροστά σε ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο. Από τη μία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πολιτιστικές παραδόσεις και τη σημαντική ε, συμβολή σε ορισμένες χώρες όπως είναι η δική μου του παιχνιδιού στην κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης του πολιτισμού και του αθλητισμού. Και από την άλλη θα πρέπει να παλέψουμε κατά της εγκληματικότητα που εγκυμονείται στα τυχερά παιχνίδια και να προστατεύσουμε του καταναλωτές ιδιαίτερα πιο ομάδες για να αποτρέψουμε τον παθολογικό εθισμό. Πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα θα πρέπει να περιτανεύσει η αρχή της ενεργού επικορικότητας που να βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ε, αρχών. Βεβαίω θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να είμαστε υπέρ της εξέλιξης ανάπτυξης κοινών ε, κανόνων και συντονισμένης ε, ρύθμισης. Ε, κατά των παράνομων φορέων εκμετάλλευσης. Επίσης θα πρέπει να εγγυηθούμε την διαφάνεια και να καταστήσουμε δυνατή μια, ένα μη διακριτικό ανταγωνισμό ο οποίος να ακολουθεί την κοινή ωφέλεια και την προστασία του καταναλωτού. Τέλος θα πρέπει να προωθήσουμε τη διαμόρφωση ενός δικτύου εθνικών οργανώσεων που να ασχολείται με τα φαινόμενα εθισμού, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων ε, και έγκαιρων πρακτικών. Κύριο Στάκουλα. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε με την Πράσινη Βίβλο στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλά αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν μπορεί να είναι λύση για το μέλλον. Θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία για να ρυθμίσουμε αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αποφύγουμε τις αντιφάσεις μεταξύ των διαφόρων προτάσεων που θα γίνουν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο τρόπος που οργανώνονται τα τυχερά παιχνίδια σε κάθε κράτος μέλος διαφέρει και ότι έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, ένα ιδιάζοντα χαρακτήρα τα τυχερά παιχνίδια. Ε, τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να πολεμήσουν τα παράνομα τυχερά παιχνίδια προφανώς, αλλά θα πρέπει και κάθε κράτος μέλος να είναι σε θέση να διαχειρίζεται αυτόν τον κλάδο και να μπορεί πραγματικά να καταπολεμήσει τα παράνομα τυχερά παιχνίδια. Θα πρέπει κυρίως να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα σε αυτόν τον κλάδο. Θα πρέπει αυτή η δραστηριότητα να γίνεται με διοντολογικό τρόπο. Και αυτό που λέει στο τέλος η έκθεση είναι απόλυτα σημαντικό. Μην το ξεχνάμε. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι κινητές επικοινωνίες ε, και η ψηφιακή επικοινωνία ε, έδωσε νέα όθηση στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Τα κράτη-μέλη φυσικά ρυθμίζουν από μόνα τους τις δικές τους αγορές, αλλά θα πρέπει να τα ρυθμίζουν με την... Αυτό θα πρέπει να γίνεται ε, σύμμορφα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Εσωτερική Αγορά. Υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν ανοιχτέ αγορές και χαμηλά επίπεδα φορολόγησης, ενώ υπάρχουν χώρες όπου απαγορεύονται τα τυχερά παιχνίδια. Ε, στις χώρες που δεν υπάρχει ε, ρυθμιζόμενη αγορά ε, τα τυχερά παιχνίδια γίνονται επιγραμμικά. Αυτό όμως έχει κινδύνους για τα παιδιά και τους εφήβους που μπορεί να αναπτύξουν διάφορες, διάφορους εθισμούς. Δεν μιλάμε για μια κλασική υπηρεσία αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Επομένως θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι ελάχιστοι κανόνες για την προστασία των ανηλίκων τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια θα πρέπει να ρυθμίζονται από αυστηρότερους κανόνες. Oui, monsieur le commissaire, nous avons obtenu... Ε, επίτροπε Πρόεδρε, Νομίζω ότι για το ΕΛΚ έχουμε ένα πολύ καλό συμβαστικό κείμενο με ελεγχόμενο τρόπο. Ανοίγουν πλέον τα τυχερά παιχνίδια. Πώ με ελεγχόμενο τρόπο θα είναι εθνική νομοθεσία και ευρωπαϊκή συνεργασία. Δηλαδή, ε, μία εφαρμογή τη αρχή Εμβέα αναγνώριση σε ένα τομέα που, σε μια αγορά που διαφέρει από όλου του άλλου, δηλαδή για την αγορά τυχερών παιχνιδιών, ενώ ταυτόχρονα τηρούμε με ενεργό τρόπο την αρχή τη επικουρικότητα, ε, δηλαδή θα έχουμε αυξημένη καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχές. Μία ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι απαραίτητη σε διάφορους τομείς. Το να γνωρίζουμε κυρίως για την καταπολέμηση της απάντησης, για την προστασία των ανηλίκων, για την καταπολέμηση των ε, παρανόμων παρόχων και την καταπολέμηση των εθισμών. Τέλος, ε, τίθε ζήτημα ακαιρεότητα στον τομέα του αθλητισμού και ελέγχου ε, των κερδών δραστηριοτήτων του τομέα αυτού. Τώρα για τους διοργανωτές των αθλητικών εκδηλώσεων Υπάρχει ένα αίτημα, ε, ε, υπάρχει ένα δικαίωμα που θα θέλαμε να κατοχυρώσουμε σε σχέση με τα στοιχήματα, τα επιγραμμικά στοιχήματα, για να αποφύγουμε την διαφθορά ε, και το παράνομο χρήμα στον τομέα αυτό. Κύριε Επίτροπε, υπερασπίζεστε μια οικονομία της αγοράς, οπότε θα πρέπει να κινηθείτε προς αυτή την κατένση. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σονάλοβα τώρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Το επιγραμμικό τυχερό παιχνίδι είναι πολύ βολικό. Ε, απλώς κάνουμε κλικ με το ποντίκι και ξεκινάει το παιχνίδι. Αλλά υπάρχει και τεράστιος κίνδυνος και κόστος για την κοινωνία. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια πολίτες, ε, το 5,5% των Ευρωπαίων πολιτών που ασχολούνται με τέτοια παιχνίδια. Ε, η προστασία από εθισμού είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνε ούτω ώστε να μην υπάρχει phishing στο ίντερνετ και προστασία των νεαρών ηλικιών, κυρίως ε, των παιδιών. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν πολύ περισσότερο σε αυτόν τον τομέα, ιδίω ε, όταν ε, καταπολεμούν αρνητικά φαινόμενα που συνδέονται με στοιχήματα και τυχερά παιχνίδια. Χαίρομαι λοιπόν που στην έκθεση υπάρχει μια έκκληση προ τα κράτη-μέλη και προ την Κομισιόν να επικεντρωθούν σε λόγου και αίτια των εθισμών, ε, ούτως ώστε να υπάρξει πρόληψη και πραγματική βοήθεια για τα θύματα του εθισμού, ε, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την αποτελεσματική καταπολέμηση των τυχερών παιχνιδιών. Ε, επιγραμμικά πάντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω θερμά αυτή την έκθεση και ευχαριστώ τον κύριο Κρόιτσμαν όλος ιδιαίτερος που ρυθμίζει, που διαχειρίστηκε πολύ ωραία μια σειρά από δύσκολε διαπραγματεύσει και ελπίζω το αποτέλεσμα θα το δεχτεί το Σώμα μεγάλη πλειοψηφία αύριο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί θα δώσουμε ένα σαφέ μήνυμα στον Επίτροπο Μπαρνιέ, που ενδιαφέρεται τα μάλλη για αυτό το θέμα, το ξέρω, για του τομεί όπου η Κομισιόν μπορεί να σημειώσει πρόοδο. Στο πλαίσιο της ενεργούς επικουρικότητας ε, και αυτή είναι μια θαυμάσια, ένας θαυμάσιος όρο προκύπτει από την έκθεση, που δεν θα υποσκάπτει την ικανότητα του κάθε κρατου μέλους να ρυθμίζει τα τυχερά παιχνίδια με βάση παραδόση και την ιστορία του, αλλά παράλληλα ε, δημιουργεί και υποχρεώσει για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, λέμε ότι αν δεν ενισχύσετε την συνεργασία σα, τότε οι καταναλωτέ δεν θα προστατευτούν σωστά σε κάθε χώρα. Και νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε ασφάλεια με όλες τις έννοιες των καταναλωτών, κυρίως των ανηλίκων, από τον εθισμό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προχωρήσουμε παράλληλα. Και νομίζω ότι χάρη σε αυτή τη δουλειά που έκανε το Κοινοβούλιο μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χάρμπορ. Στο τελευταίο ομιλητή και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές, εδώ και 18 μήνες δεσμεύτηκα ενώπιόν σας να ξεκινήσω μια πλατιά διαβούλευση για το θέμα αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό για τα τυχερά παιχνίδια online. Και σήμερα λοιπόν επανερχόμαστε στο θέμα αυτό και θα ήθελα εγώ από την πλευρά μου να επανέλθω υποδηλώνοντας την ε, στεναρή μου πρόθεση να μεταφράσω ε, και να μεταφέρω πέρα από αυτή τη διαβούλευση τα βασικά συμπεράσματα στην πράξη. Έλαβα πάνω από 250 απαντήσεις ε, σε σύνδεση με τα πέντε ατελέ εμπειρογνωμόνων σε σύνδεση με τις ε, εντατικές συζητήσεις που κάνατε εσείς για την έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Κρότσμαν. Και όλα αυτά δηλώνουν ξεκάθαρα αυτό το δυναμισμό υπέρ μιας συγκεκριμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την δημιουργία ενός βασικού ε, ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο να σέβεται, όπως είπε ο κύριος ε, Χάρμπουρ, την, αρχή της ενεργού επικαιρικότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρότσμαν για τη δέσμευσή του, αλλά επίσης την κυρία Σάλ Μόζε, την κυρία Ρούλε, τον κύριο Αμπάντ, τον κύριο Τεζόν και τον κύριο Φόξ για τις εισφορές τους σε αυτή την έκθεση η οποία ε, δείχνει μια μεγάλη σύγκληση απόψεων και συμφωνίες προς τη διάγνωση. Δηλαδή στο online περιβάλλον καμία χώρα μέλος δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει από μόνη της την προστασία των καταναλωτών και των πολιτών και ε, ε, αυτά στηρίζουν τα όσα είπε ο κύριος Ντάλι εν γέννη ε, για την προστασία των καταναλωτών. Δεύτερον, οι καταναλωτέ και το σύνολο των πολιτών θα πρέπει να μπορούν να υπολογίσουν μια ελάχιστη προστασία η οποία να είναι ίση και αποτελεσματική, ιδιαιτέρω για του νέου και του ανηλίκου όπω ε, επεσήμανε προηγουμένω η κυρία Ρόιτεβα. Και αυτά ανεξάρτητα από την πλατφόρμα παιχνιδιού που παίζουν. Τρίτον, εάν κάθε χώρα μέλο παραμένει ελεύθερη να ορίσει το εύρο ανοίγματο τη αγορά σεβόμενη την ε, αρχή τη συνοχή, ε, είναι ξεκάθαρο ότι κατευθυνόμεθα προς, ένα μέτριο παθές άνοιγμα πολλών αγορών ε, ελήψη ε, νόμιμης προσφοράς στην Ευρώπη οι Ευρωπαίοι πολίτες παίζουν σε παράνομους ιστότοπους τρίτων χωρών που δεν είναι προστατευμένοι και εξυπηρετούν το ξέπλυμα χρήματος. Πέμπτον, θα πρέπει να επαγρυπνήσουμε ούτως ώστε να προσφέρουμε ελκυστικές προϋποθέσεις φορείς εκμετάλλευση των τυχερών παιχνιδιών online αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους παίκτες και να καταπολεμήσουμε την απάτη. Έκτον, θα πρέπει να δράσουμε γιατί το μέσο αυτός βρίσκεται σε πλήρη επέκταση. Έχει ένα τζίρο 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 και μπορεί να φτάσει στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 και έστω και αν αυτό αντιπροσωπεύει 14% της αγοράς των παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 45% της παγκόσμιας αγοράς των online παιχνιδιών και θα πρέπει λοιπόν να συνοδεύσουμε τον τομέα αυτό στην επέκτασή του επαγρυπτώντας για την επαρκή του πλαισίωση. Ποια θα έπρεπε να είναι λοιπόν, ποιος θα έπρεπε να είναι ο δικός μας χάρτης για να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις μας, σε όλες τις δικές ερωτήσεις και σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξεκάθαροι. Η εναρμόνιση δεν ε, βρίσκεται στην μερίσια διάταξη, ωστόσο κάποιε κοινέ δράσει, ορισμένα θέματα κλειδί μπορούν να εξεταστούν και χωρί αμφιβολία στο τέλο του δρόμου αυτού θα υπάρξει ένα βασικό πλαίσιο κοινή ρύθμιση. Ε, θα ήθελα να αναφέρω δύο ή τρία θέματα κλειδί επί των οποίων θα πρέπει να δράσουμε. Πρώτον, τον διάλογο μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα συνεργασίας μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών που απορρέουν από μια έλλειψη αμοιβέ εμπιστοσύνη, πέρα από ορισμένε διμερεί συμφωνίε και μια πρόσφατη απόπειρα να δημιουργεί μια κοινή πλατφόρμα, δεν υπάρχει μια κουλτούρα συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Αντιθέτω, παρατήρησα ότι συχνά υπάρχει σημαντική έλλειψη εμπιστοσύνη. Χωρί όμω έναν νέο. Χωρί όμω μια αύξηση αμοιβαία εμπιστοσύνη, δεν είναι δυνατόν να σημειωθεί καμία πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ενίσχυση των ελέγχων και την προστασία των παικτών, ιδιαίτερα των νέων. Η προτεραιότητα θα πρέπει λοιπόν να δοθεί σε αυτή την συνεργασία των, ευρωπαϊκών, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Δεύτερο στοιχείο κλειδί μία ελάχιστη απέτηση, ελάχιστο κατόφλι προστασία. Θα πρέπει να εγγυηθούμε σε όλους τους Ευρωπαίου προστασίες, ε, Ευρωπαίους πολίτες συγγνώμη, ένα επίπεδο προστασία και πρωτίστω του νέους. Θα πρέπει να ε, υπάρξει μια επαγγελματική συνεργασία των τυχερών παιχνιδιών που σήμερα αυτορυθμίζονται ε, και εφαρμόζονται διάφορες ε, προδιαγραφές. υπάρχει λοιπόν Μία έκκληση την οποία απευθύνετε κι εσείς ε, κύριε Κρόιτσμαν προς την κατεύθυνση μιας νομικής ε, σαφήνειας. Τώρα, η καταπολέμηση της απάτης. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη συνένεση στο πλαίσιο αυτής της διαφούλευσης και σε αυτά που λέτε εσείς. Στο σύνολο των επιγραμμικών τυχερών παιχνιδιών όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας κατά του ξεπλήματος χρήματος που αυτή τη στιγμή καλύπτει μόνο τα καζίνο. Θα ήταν σημαντική λοιπόν ο πρόεδρος στην κατεύθυνση της πλαισίωσης του τομέα αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέμπτο θέμα κλειδί είναι η ανεξαρτησία. Η κυρία, κυρία η κυρία Σανέλαβα το ανέφεραν προηγουμένω, δεν είναι δεδομένο να μιλούμε σοβαρά για την προστασία των καταναλωτών χωρί την αναγνώριση τη ανάγκη διεξαγωγή ερευνών για τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία συνδέονται με τα παιχνίδια και τα φαινόμενα εξάρτηση. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τι δυνατότητε έρευνά μα για ένα θέμα που ορισμένε φορέ θεωρείται περιθωριακό, αλλά εγώ δεν θεωρώ καθόλου περιθωριακό ή ελάσσον. Τώρα, η ακαιρεότητα του αθλητισμού είναι το πέμπτο θέμα κλειδί. Και εδώ, κύριε Κρό, Κυρίε κυρίες και κύριοι, ε, θα πρέπει να ε, επαγνυπνήσουμε για τα θέματα αθλητικής απάτης και θέλουμε να δώσουμε αποτελεσματικέ λύσει. Μία την ιδέα ενό ευρωπαϊκού ορισμού της αθλητική απάτης και μιας ε, ποινικοποίηση αυτού του φαινομένου. Ενδιαφέρουσα ιδέα. Είναι δύσκολο βεβαίω να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να το προσεγγίσουμε το θέμα αυτό αυτοσχεδιάζοντα. Χρειάζεται να προηγηθεί τεχνικό και νομικό έργο και η ιδέα μου είναι να συνεργαστούμε με συναδέλφου που ενδιαφέρονται άμεσα, τον κύριο Βασιλείου, την κυρία Ρέντινγκ και τον κύριο Νταλή από την πλευρά των καταναλωτών. Είμαι πεπισμένο ότι ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιοι πρόοδοι για μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ αθλητικών ε, ενώσεων, ε, μεταξύ των φορέων εκμετάλλευση και των ρυθμιστικών αρχών, ούτω ώστε να αποτρέψουμε το στήσιμο ορισμένων αγώνων. Έκτον, ε, η συμβατότητα των ε, εθνικών ε, νομοθεσιών με τη συνθήκη. Ο κύριος Τακούλα αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, γιατί αναφέρθηκε ο ίδιος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που είναι ξεκάθαρο όσον αφορά του περιορισμούς που μπορούν να δικαιολογηθούν υπέρ του κοινού συμφέροντο. Θεωρώ κύριε Τακούλα ότι στο τομέα αυτό για να προχωρήσουμε θα πρέπει να υπάρξει μια σαφήνεια εν σχέση με αυτό το οποίο διαφοροποιεί μία παράνομη από μία νόμιμη ε, προσφορά, το οποίο, θέμα το οποίο θέτει συμβατότητα των εθνικών νομοθεσιών με την ε, συνθήκη. Πώς τώρα, ξεκινώντας από αυτά τα θέματα κλειδιά και ξεκινώντας από τις ε, δικές σας προτάσεις, κύριε Κρότσμαν, θα εργαστούμε. Ε, σε μια πρώτη φάση θα κινηθούμε προς την ε, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και έχω την πρόθεση τις επόμενες εβδομάδες να ανοίξω ο ίδιος μια συνάντηση όλων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη το οποίο μέχρι στιγμή δεν υπάρχει, ούτω ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις αυτής της συνεργασίας. Επίσης όπως, ε, καθώς η συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αναχών μας επιτρέπει μια πρόοδο σε αυτά τα θέματα κλειδί που αναφέρατε εσείς αλλά και ανέφερα και εγώ, ε, κυρίως κάτω από το πρίσμα της ανάγκης συμπληρωματικών δράσεων θα εργαστούμε σε μια δεύτερη φάση η οποία θα μπορούσε, όπως ζήτησε ο κύριος ε, Πάσκα, να στηριχθεί σε ρυθμιστικές πρωτοβουλίες κλειδί όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές, τις ελάχιστους κανόνες. Εδώ θα είμαι ιδιαίτερος ξεκάθαρος, είμαι μέλος ενός σώματος και θα πρέπει να συνεργαστώ με όλους τους στο πλαίσιο αυτό, ούτως ώστε να συμμεριστούμε όλη αυτή την πεποίθηση. Ε, ε εργαζόμαστε λοιπόν ως ρυθμιστές και στη βάση αυτής της πρώτης διαπίστωσης, του πρώτου έργου, θα ήθελα να συμμεριστώ με τους συναδέλφους την πεποίθηση να πάμε πιο μακριά όσον αφορά τη δημιουργία μιας ελάχιστης ρυθμιστικής πρωτοβουλίας. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε την διαδοχή των φάσεων, τη μία μετά την άλλη. Ε, ανέφερα τα βασικά διακυβεύματα και τώρα θα ήθελα να πω θα εργαστώ κάτω από το πρίσμα της δικής έκθεσης κύριε Κρόιτσμαν και η πρόθεσή μου είναι μετά από τις διαβουλεύσεις του σώματος να σε υποβάλω ένα συγκεκριμένο πλάνο δράση το οποίο θα υποβάλω στο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κατά τα μέσα του 2012. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρόιτσμαν, σας ευχαριστώ πολύ κύριοι βουλευτές για αυτή την έκθεση η οποία θα διευκολύνει το έργο της Επιτροπής στο μέλλον. Έχουμε μια συλλογική ευθύνη και οι χώρε μέλη να ρυθμίσουν τα παιχνίδια αυτά, να προστατεύσουν του καταναλωτέ, ιδιαίτερω τους ανηλίκους, να καταπολεμήσουν την απάτη και ε, να αναπτύξουν μια επαρκή συνεργασία. Θα ήθελα να σας διαβεώσω για την δική μου στεναρή πεποίθηση όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα και τη δέσμευση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρνιέ. Ε, κύριε συνάδελφε, έχει κλείσει η συζήτηση και θα γίνει η ψηφοφορία αύριο στις 12 για το θέμα αυτών των τυχερών παιχνιδιών online. Τώρα θα συζητήσουμε για τη μελισσοκομεία.